Bien, mes chers collègues, je vous invite. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σα. Κηρύσω την έναρξη τη έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή των Προπολογισμών. εξετάζουμε αν έχει εγκριθεί η σε διάταξη, δεν έχετε τηρήσεις. Προτείνω επίσης τα πρακτικά του τριμερούς διαλόγου που είχε θετική κατάληξη σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να υποβληθούν στο τέλος της συνεδριασέως μας και ευκρινίζω ότι στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται ένα επιπλέον σημείο για τις μεταφορές. Η κυρία Χολμάιερ θα μας κάνει σχετική παρουσία στο σημείο c 5. Άρα έχουμε να συζητήσουμε εντολή εν ώψη διαπραγματεύσεως για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό 2016. Η Επιτροπή μέσω της κυρίας Γεωργίευα μας υπέβαλε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016 και δίνω τον λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες ώστε να μας παρουσιάσει το πώς αναλύει και ποιες είναι οι κύριες γραμμές αυτής της αντολής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας τα πω στα Έχουμε σαφείς ε, κατευθυντήρες ε, που υιοθετήθηκαν στην Ολομέλεια. Σας υπενθυμίζω ότι τα τρία e η, τα αγγλικά ε, οι επιχειρήσεις, το επιχειρήν και η ε, απασχόληση και όταν μιλάμε για επιχειρήσεις κυρίως μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η βασική ε, κατεύθυνση του προπολογισμού. Πρόκειται για το τομέα 1α. Επίσης όμως μας ενδιαφέρει και η εσωτερική συνοχή, ε, αλληλεγγύη. Και σε αυτό το πλαίσιο μην ξεχνάμε την πολιτική συνοχής που επίσης βοηθάει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και επίσης και την εξωτερική αλληλεγγύη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος πάρχος ε, δωρεάν βοήθεια στον κόσμο. Ε, η συνολική παρουσία της Ευρώπης στον κόσμο μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πολύ σημαντική. Όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονία μας ε, καλύπτονται από μηχανισμούς ε, που εκφράζουν την εξωτερική μας αλληλεγγύη. Πρόκειται για τον τομέα 3 και τον τομέα 4 που είναι επίση πολύ σημαντική. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την πρόταση της ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη μια έκθεση, ένα προσχέδιο έκθεσης για εντολή. Να χαιρετήσω την πρόταση της Κομισιόν και ε, να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που πρέπει να είναι σαφής. Πρόσφατα έγινε με επιτυχία διαπραγματεύση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα συνεχίσουμε όμως με στόχο την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου επί του ε, προγράμματος Ορίζοντα 2020 και επί του μηχανισμού ε, του χρηματοδοτικού μέσου σύνοντας στην Ευρώπη. Και θα υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο αυτό που είχε αγνοηθεί ότι για να ε, ε επικυρωθεί το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, το κοινοβούλιο είχε απαιτήσει και έγινε δεκτό να, ε, να εφαρμόζεται η αρχή της ευελιξίας και το σχέδιο Juncker για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε περιθώρια τα οποία είχαμε και το Συμβούλιο είχε ξεχάσει την ύπαρξη αυτών των περιθώριων. Αυτό, το, αυτά τα περιθώρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς. Εμείς θέλουμε έναν ε, προπολογισμό αποτελεσματικό. Αυτά τα περιθώρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις προτεραιότητες μας, για πολιτικούς λόγους δηλαδή, για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ιδιαίτερος για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, που είναι μία από τις προτεραιότητες μας. Το κόσμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούσε ε, προτεραιότητά μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ε, έχει ε, τις ε, ε, πιστώσεις υποχρεώσεων να αυξάνονται συγγνώμη, δεν, ε, δεν βλέπει αύξηση, κάτι που δεν συμβαδίζει με τις ε, προτεραιότητές μας. Για την απασχόληση των νέων το 2016 ε, δεν έχουμε ανάληψη υποχρεώσεων εξαιτίας του front loading, οπότε θα πρέπει να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε δηλαδή γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο. Να έχουμε μια τεράστια ενεργεία νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε πόρους, κονδύλια και να μην μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Είναι σημαντικό τα κονδύλια που διαθέτουμε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ε, ως γενικό σχόλιο επίσης να πω και το εξής. Η αρχή μας είναι <clears throat> ότι η ανάληψη υποχρεώσεων ή, ή, ή, ή θα, τύχουν σεβασμού. Και τι εννοούμε. Ε, η, η ευελιξία είναι μία δέσμευση. Αλλά και όλα τα προγράμματα, η πολιτική στόχη του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος ε, πλαισίου ε, θα πρέπει να εκτελούνται κανονικά έτσι ώστε να μην υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη που θα πρέπει να αισθάνονται οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν απαράδεκτο εμείς να μην τροφοδοτήσουμε αυτά τα προγράμματα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, για τα οποία έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις με τα κατάλληλα κονδύλια. Θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών το οποίο ε, συμφωνήθηκε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ε, έχουμε πια βαρεθεί να μιλάμε για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι μέσα στην καθημερινότητα και όχι κάτι έκτακτο. Ε, δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε πιστώσεις και στο τέλος να μην εκταμιεύονται τα ποσά. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί. Χαιρέτησα λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν για τον προπολογισμό 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, σε, αν, σε αναλήψεις ε, ε, πιστώσεων και 143,5 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 2,4% σε αναλήψεις πιστώσεων και 1,6% σε πιστώσεις πληρωμών. Υπάρχει και ένα περιθώριο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις πιστώσεων και από αυτά τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 1,2 είναι στον τομέα 2 υπάρχει και κάτι άλλο θετικό που είναι η μα και αρνητικό ταυτόχρονα η χρήση στον τομέα 3 όλου του περιθωρίου Δηλαδή χρησιμοποιούμε το σύνολο της ευελιξίας που μας δίνεται. Ε, εμείς ε, έχουμε ως αρχή ότι ο μηχανισμός ευελιξίας ε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι απαραίτητο. Διότι υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να μας οδηγούν στο να ξεπερνάμε τα ανώτατα όρια. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε τα περιθώρια να διατηρούνται. Σε ό,τι αφορά τον καθένα από τους τομείς, τομέας 1α, έχουμε αύξηση στην άλυψη πιστώσεων κατά 6,1% και σε πληρωμές 11,4%. Σε αυτό τον τομέα είναι προφανές και όπως το έχουμε πει επανειλημμένως θα ε, περιλάβουμε το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων το μηχανισμό χρηματοδοτικό μηχανισμό σύνδοντας στην Ευρώπη και εκεί θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού ε, να επιστρέψουμε αυτό το οποίο είχαμε αποσύρει από αυτό το μηχανισμό για τη δημιουργία του Ταμείου. Ε, θα πρέπει, όπως έχουμε πει, να τυχαίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις μας ε, και πρέπει να γίνουν σεβαστές και στο Ταμείο και στον χρηματοδοτικό μηχανισμό συνέντας στην Ευρώπη. Το <clears throat> Κοινοβούλιο δεν πρέπει να είναι μόνο του σε αυτόν τον αγώνα. Θα πρέπει να βοηθηθεί από την Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν διαχειρίζεται αυτά τα προγράμματα. Και βέβαια και το Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του και τι δεσμεύσει, να τηρήσει τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Στην, στον τομέα 1β έχουμε αύξηση 3,2% σε σχέση με το 2015 στις ε, πιστώσεις ε, ανάλυσης υποχρεώσεων και μια μείωση στη πιστώσεις πληρωμών, μείωση κατά 4%. Και θα πρέπει να δούμε μήπως αυτό ε, αμφισβητητό συμβιβασμό Ε, έχουμε μια υστέρηση κατά 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα έτη 2007-2013 πληρωμές. Θα πρέπει να δούμε αν ο συμβασμό που βρήκαμε, ε, που στον οποίο είχαμε καταλήξει, αμφισβητείται από αυτή τη μείωση των πληρωμών. Και θα πρέπει να δούμε και την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ε, που όπως σας είπα δεν ε, έχει πιστώσεις το 2016 και πρέπει να δούμε πώς, τι θα γίνει. Τομέας 2 και εδώ έχουμε μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2015 στις ε, πιστώσεις σε ανάλυση υποχρεώσεων και στις πληρωμές. Μείον 0,1%, μείον 0,2% αντίστοιχα. Ε, <coughs> περιμένουμε βέβαια το ε, την ε, τροποποιητική επιστολή της Επιτροπής ε, τον Οκτώβριο για να δούμε τη συνέχεια. Εδώ έχουμε κάποιες αυξήσεις σε προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται και αυτό είναι καλό. Μήμα 3, εδώ δεν θα έχουμε περιθώριο. Χρησιμοποιείται δηλαδή ο μηχανισμός ευελιξίας καθ' 127 εκατομμύρια ευρώ Εδώ έχουμε τα σχέδια, τα πιλωτικά σχέδια και τις ε, δράσεις προετοιμασίας που θα πρέπει να συνεχιστούν. Σε ό,τι αφορά τον τομέα 4 που θα πρέπει να τη διαβάσουμε παράλληλα με, με τον τομέα 3 ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Χαιρετίζουμε την αύξηση που προτείνεται ε, στις πιστώσεις άναληψης υποχρεώσεων 5,6% και το θέμα της αύξησης κατά 28,5% των πιστώσεων πληρωμών. Ε, πρέπει όμως να σχετικοποιήσω αυτό που είπα μόλις τώρα, γιατί αυτές οι αυξήσεις γίνονται χάρη στις ε, ε, πληρωμών του παρελθόντος. Και είναι ντροπή που χρειάζεται να πληρώσουμε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως ε, τόκους υπερημερίας για πληρωμές που δεν είχαν γίνει ε, το 2005 στον τομέα 4. Πρόκειται για καθυστερήσεις πληρωμών οι οποίες κοστίζουν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται κάθε χρόνο. Ε, που όμως ε, σίγουρα δεν αμφισβητεί τις προτεραιότητες που έχουμε. Οι πληρωμές δηλαδή, το θέμα των πληρωμών των, ε, που υστερούν θα πρέπει να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από τις προτεραιότητες μας, χωρίς να θυγούν αυτές. Σε ό,τι αφορά τα, σχέδια, τα σχέδια, το είπα, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τα ποσά τα οποία είχαμε πει. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, τομέας 5, χρειάζεται λιτότητα, αυστηρότητα, έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ελάχιστο διοίκησης και διοικητικής ισχύω έτσι ώστε να φέρει σε πέρα τι υποχρεώσει τη. Ελπίζω ότι αυτέ οι γενικέ γραμμέ προσανατολισμού θα βοηθήσουν το Συμβούλιο να ε, κάνει μια καλή ανάγνωση τη πρόταση του κανονισμού όπως προτάθηκε, ε, του προπολογισμού όπως προτάθηκε από την Κομισιόν ε, στις 23 Ιουνίου ε, στην Επιτροπή εμείς εδώ ε, τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια 14 Ιουλίου έχουμε τριμερή διάλογο και περιμένουμε από το Συμβούλιο μια συμβαστική και επικοδομητική στάση, μια στάση που θα ε, σέβεται τις ε, παλαιότερες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και βέβαια το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Je remercie Ευχαριστούμε τον και Μπράβο του που ασχολείται με τόση ζέση με το θέμα και επίσης είναι εισηγητής και όσον αφορά την νομική πτυχή του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ, και επίσης ε, εκπονεί και την ε, έκθεση αυτή σε σχέση με την ε, εντολή για να καλυφθεί και τον ευχαριστούμε. Οπότε που θα ε, μιλάμε για ανάπτυξη, να στρέψουμε το ρήμα για την ανεργία, να καταπολεμήσουμε το σκάνδαλο της ενεργείας των νέων στην Ευρώπη και στη συνέχεια να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε ε, τις μεταναστευτικές ροές. Είναι οι προτεραιότητες που ελπίζουμε ότι θα καλυφθούν από τον προπολισμό του 2016. Και τώρα αρχίζουμε την συζήτηση. Αλλά και ε, αν θέλουμε να λάβει το λόγο και η Γενική Συγκεκριτή του Πρωθυπουργού, κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίως και θα επιστρέψουμε στις λεπτομέρειες και εγώ θα σας πω απλώ όμως ε, κάποιες γενικές παρατηρήσεις γιατί σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με την εντολή που αφορά τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφές ότι ο βασμός του 2016 θα είναι και πάλι ένας τέτοιος προϋπολογισμός που θα καλύψει τις προτεραιότητες του μέλλοντος και όχι ε, τα ανεξόφλητα του παρελθόντος. Άλλωστε έχουμε και τα εθνικά στοιχεία του 2015 όπου έχουμε αυτά τα 20 δις ανεξόφλητα και το 2016 επομένως τουλάχιστον αυτό θα εξοβαλυνθεί και επομένως έτσι θα ενατενίσουμε το μέλλον. Επίσης η συζήτηση το 2016 θα μας ε, ωφελήσει ώστε να ε, βρει συνέχεια αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Βερνάντης για την διαπραγμάτευση για τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση ε, του, του δημοσιονομικού πλαισίου γιατί έχουμε αυτές τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να τις σχετιστούμε όπως το ΕΦΣΙ της Επιτροπής Γιούγκερ, αλλά έχουμε επίση και την πρόκληση της Μεσογείου. Έχουμε την μεταναστευτική κρίση, έχουμε τις μετακινήσεις των προσφύγων, έχουμε την κατάσταση στην Ουκρανία, τις σχέσεις με τη Ρωσία, πολλά νέα στοιχεία τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί. Αλλά λογικό είναι αυτό, δεν καλύπτονται από αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε και αυτά θα περιληφθούν ε, στην συζήτηση και επομένως θα πρέπει να αναλύσουμε για το 2016 τον προϋπολογισμό σίγουρα αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θέλουμε να προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου γιατί έχουμε αυτές τις προτεραιότητες που θα πρέπει να καλυφθούν δεν καλύπτονται από τα στοιχεία προβλήματα τώρα, από τα ποσά τώρα, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει για όλε αυτέ τι προτεραιότητε που τη βρίσκουν σύμφωνοι. Αλλά όπω είπα στην αρχή, ε, οι σοσιαλιστές πρόκειται να επεξεργαστούμε στις λεπτομέρειες του. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Και Γίτσες, αγαπητοί συνάδελφοι. Εσείς. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Φερνάντας Γενικό Εισηγητή για την ε, πολύ καλή έκθεση και τη δουλειά που έχει κάνει. Εκ μέρου της μου θέλω να πω ότι μπορώ αφενός μένα να δεχθώ πολλά από αυτά που είπε. Βεβαίως και έχουμε και εμείς ε, ακούσει θέματα σχετικά με τις προτεραιότητες στο χώρο, στον τρόπο εργασίας μας για θέματα που δεν είναι αμφισβητούμενα. Τα εξωτερικά σύνορα, την διασφάλιση τους, αλλά και την προσφορά βοήθειας ε, σε εκείνους που κινδυνεύουν από πνιγμό μέσα στη Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν αδιαφιλονίκη τα ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως λέμε και ότι θα πρέπει και στον προπολογισμό 2016 να ε, τηρήσουμε τις κύριες γραμμές μας, να μην τις λησμονήσουμε και να κάνουμε τις επιλογές για το τι είδους πολιτική θέλουμε. Ιδιαίτερα στο τομέα του προπολογισμού λοιπόν θέλουμε περισσότερη επικουρικότητα δεν θέλουμε εξάπαντος να υπάρχει μια συλλήβδην γενική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για όλα τα θέματα. Θέλουμε να κοιτάμε προσεκτικά πού πάνε τα χρήματα, για ποιο λόγο διατίθενται τα συγκεκριμένα κονδύλια και εάν στον τομέα για τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια πρέπει να έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δραστηριοποιείται. Και για να μην σας καθυστερήσω άλλο, έχουμε δύο πτυχές πολύ σημαντικές. Όσα πολύ σημαντικές αξιολογήσει. τις έχουμε συζητήσει αρκετές φορές νομίζω, ένα ζήτημα με τους μη εξοφλημένους λογαριασμούς, όπου για να είμαστε σοβαροί, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να κοιτάξουμε, να θέσουμε το ζήτημα αυτό ως κύρια προτεραιότητα της εντολής. Και νομίζω ότι μόνο εάν δεν επιτρέψουμε την απεριόριστη αύξηση των πιστωσών ανάληψης υποχρεώσεων ε, μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να συγκρατήσουμε το πρόβλημα. Φαίνεται όμως τώρα ο κ. Φεράντας να προτείνει κάτι διαφορετικό και βεβαίως έχουμε ακούσει πολλά ωραία και από την κυρία Κεωργίευα την Επίτροπο αλλά ε, είναι άλλο πράγμα να ενισχύουμε τα ποσά αυτά και άλλο να νομίζουμε ότι μπορούν να υλοποιηθούν κιόλα. Επίσης, το τρίγωνο Επιτροπή Συμβούλιο Κοινοβούλιο το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να εξαντλεί την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου σε μια φαινομενική mm. εκπροσώπηση δηλαδή θα πρέπει να μπορούμε και σε σχέση με τα έσοδα να έχουμε λόγο και στην απόφαση. Ωστόσο αυτό είναι στα χέρια των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει το Συμβούλιο πλέον να συμπεριφέρεται σαν να μπορούμε και εμείς στο Κοινοβούλιο δηλαδή να επηρεάζουμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις για τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον το ορίζουμε οι συνθήκες λοιπόν πρέπει και εμείς να είμαστε θέση να λέμε ότι όποιος ε, δίνει την έγκριση για μία δαπάνη πρέπει να είναι σε θέση να βρει και την χρηματοδότησή της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλή. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάνδες για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση μας ανέλησε λεπτομερώς τις ε, διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού. Εμείς βλέπουμε να προσδιορίζονται και να ακολουθούνται κύριες εταιρεότητε από τον προπολογισμό αυτών, δηλαδή απασχόληση, επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη. Οι πιστώσεις πληρωμών ενισχύονται κατά 1,5%, οι εραλήψεις υποχρεώσεων κατά 5,5%. Στα τέλη του 2016 αναμένεται Και πρέπει να πω ότι το έχουμε συστήσει εδώ πλειστάκες. Έως το τέλος λοιπόν του 2016 θα έχουμε πιστεύω εξασφαλίσει τη μείωση των ραλ των υπόλοιπων προς ε, ρευστοποίηση και ότι θα υπάρχει υποστήριξη για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και μέτρα για την εκπαίδευση, για την καινοτομία, την έρευνα ότι θα έχουμε κονδύλια για το Ταμείο Εγγύησεων για την γεωργία και τους γεωργούς και ότι θα υπάρξει επιπλέον υποστήριξη με κονδύλια για τα θέματα της μετανάστευσης. Εδώ λοιπόν θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της εξωτερικής διάστασης της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα λοιπόν η αύξηση στις πιστώσεις των πληρωμών παρακολουθεί πρέπει να σημειώσουμε τον πληθωρισμό άρα σημαντική αύξηση δεν βλέπουμε παραμένει στα ίδια επίπεδα δηλαδή ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης με το προηγούμενο έτος Κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε στην πολιτική της συνοχής γιατί μιλάμε για οικονομική και κοινωνική συνοχή βλέπουμε να μειώνεται κατά 4% η χρηματοδότηση. Σε μια περίοδο όμως όπου αυξάνεται όλο και περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν νομίζω ότι στον τομέα αυτών ειδικά πρέπει να γίνονται περικοπές. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι πιστώσεις πληρωμών για τη διοίκηση οι οποίες ξαρώνται κατά 3%. Ελπίζω να έχει γίνει πολύ προσεκτικός υπολογισμός. Εμεί γενικά υποστηρίζουμε τον προϋπολογισμό στα θέματα της καλύτερης επασχόλησης, της αντιμετώπισης της μετανάστευσης, της αντιμετώπισης των ε, της παγκοσμιοποίησης και όλων αυτών των ζητημάτων και ελπίζουμε ότι τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να τις προασπίσουμε κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ευχαριστώ. Κυρία Νίριαντα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον εισηγητή για την λεπτομερέστατη αυτή ε, ανάλυση της κατάστασης θα συμπληρώσω δεν θα, επαναλάβω αυτά που υπόθηκα νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερα στις παρατηρήσεις να τονίσετε το ζήτημα της απασχόλησης και της δημιουργίας της θέσεων καθώς μάλλον στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο δεν υπάρχουν επιστώσεις ε, ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με, με τη δημιουργία θέσεων εργασία και τα ζητήματα κόσμε και οτιδήποτε έχει σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιπλέον έχουν περικοπεί. Πρέπει λοιπόν τις προτεραιότητες να τις ορίσουμε εκεί που είναι οι πραγματικές ανάγκες, δηλαδή στην αξιοπρεπή απασχόληση της θέσης εργασίας. Ιδιαίτερα στο θέμα της μετανάστευσης θέλω να σταθώ για να πω ότι πρόκειται για ένα κεντρική σημασία θέμα, ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Η εστίαση και προτεραιότητες είναι σε λάθος σειρά νομίζω. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τα πρώτα καταλήματα και υποδοχή αλλά και την ενσωμάτωση στις κοινωνίες και πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά επίσης το πώς μπορούμε να ε, την τους αυτή πληγή που είναι ε, οι χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να μένουν οι πολίτες εκεί και που χρειάζεται να βοηθήσουμε με μέτρα ε, υπέρ της ειρήνης κτλ. Το ζήτημα επίσης του μικρού περιθωρίου που έχουμε στις κύριους τίτλους του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει πολύ σαφή τοποθετήσεις σε σχέση με το πολιτές νομικό πλαίσιο και τον όλο του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον για γιατί εξαντλητικά διεξήλθε την έκθεση για όσα θα κάνει και επίση να προσθέσουμε και κάποια ζητήματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δείξει πρώτα-πρώτα. Η πολιτική μα ομάδα θεωρεί ότι από την του 2017 δεν είναι δυνατόν να μην καλύπτουμε τι πιστώσει του 2016. Θα πρέπει να κάτσουμε και να προβληματιστούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των πόρων. Γιατί προς τα γη κινούμεθα. Και συνέχεια θα δούμε πώς θα το διαρθρώσουν αυτό και να δούμε πώς η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στο performance budgeting. Και κατόπιν, επίσης πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ για τις προτεραιότητες όπως τις ανέφερε ο συνάδελφος πριν από λίγες μέρες είχαμε μια διάσκεψη στο Τρέντο, είχαμε μια διεθνή έκθεση και εκεί ήρθαν κάποιοι διεθνεί ε, οικονομολόγοι βραβευμένοι με ε, Νόμπελ όπω ο Κρούγμαν και ο Στίγλιτς και συζητήσαμε για την ανάπτυξη, για τις ανισότητες και ε, ιδίως για συζητήσαμε το τι γίνεται στις αναπτυγμένε βιομηχανίες όπως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα φροντίσουμε εκείνα τα κονδύλια τα οποία βοηθούν να συρρυκνωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών αυτές πώς θα καλυφθούν και πώς αυτές θα καταστούν μια προτεραιότητα. Τώρα για τις λοιπές προτεραιότητες. Ε, βέβαια και συμφωνούμε για τις επενδύσεις. Για τη διαχείριση των μεταστηρικών ροών για το πρόβλημα της ανεργίας. Θέλουμε με θάρρος να γίνει καλύτερη αξιολόγηση και να δούμε τι περικοπές μπορούν να γίνουν στο νούμερο 4 όσον αφορά το Global Europe. Και να δούμε αν χρειάζεται σήμερα το πρόγραμμα αυτό, αφού γιατί σήμερα θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και τους διαθέσιμους πόρους στο ιστορικό των 28 κατά το μέλλον. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με ε, τα άλλα προγράμματα, τα άλλα μέσα και να δούμε πώς μπορούμε αυτά να τα αναδιαρθρώσουμε όταν γίνει η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Τελευταίο τώρα, κατάσταση των πληρωμών. Παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη διαδρομή που έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτάσεις. Και από δική μας πλευράς ακόμη υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δράση για το διευθυντικό πρόβλημα. Δηλαδή να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των υποχρεώσεων και πληρωμών σε παρόμοια επίπεδα. Και να προβληματιστούμε επίσης για το πώς θα έχουμε περισσότερη επικουρικότητα στον ε, προϋπολογισμό. Να κάτσουμε δηλαδή και να αξιολογήσουμε τον σημερινό μηχανισμό του προϋπολογισμού που η Ευρώπη σήμερα είναι η θέση να κατανείμει στα κράτη-μέλη τους πόρους που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την βελτίωση του δυτικού επίπεδου των Ευρωπαίων. Να μια σκέψη τώρα. Όσον αφορά τη μετανάστευση, να σας επισημάνω ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού ανέλησαν μια μελέτη η οποία θα αφορά τους πόρους τους σχετικούς με την μετανάστευση. Θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αρχές Ιουλίου καθώς και κάποιες σχετικές συστάσεις. Οπότε τότε θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής μας να ρίξουν μια ματιά σε αυτά και να δούμε τι θα γίνει με τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Γκάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως και ο του κυρίου Φερνάντες δεν έχω να πω πολλά επικριτικά σε σχέση με την παρουσίασή του. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Ε, μας έχει περιγράψει ικανοποιητικά τις διάφορες κατηγορίες των δαπανών ακολουθεί την πολιτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις επιλογές ίσως ένα-δύο σημεία λεπτομέρειας να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε με μικρές τροπολογίες. Είχα παραδείγματι την εντύπωση πως θα έπρεπε να μας απασχολήσει κάπως περισσότερο εάν δεδομένη της κρίσης πληρωμών Πρέπει να συνεργαστούν τα θεσμικά όργανα ώστε οι πληρωμές να ακολουθούν πιο κοντά, πιο προσεκτικά τις δεσμεύσεις ανάληψης, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Και όπως είπε ο κύριος Κέμε, εγώ θα πρότεινα και το αντίστροφο να γίνει, δηλαδή να προσέξουμε βεβαίως να μην αναλαμβάνουμε υπερβολικά υψηλές ε, υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και τις πιστώσεις των πληρωμών εκεί που έχουμε αναλάβει ήδη τις υποχρεώσεις. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη και έχουμε ορίσει πολιτικές επιλογές οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη σε συνεργασία και με την ε, συμφωνία του Συμβουλίου. Όλα αυτά χρόνια λοιπόν υπάρχει μια πολιτική τοποθέτηση, αναλαμβάνει το Συμβούλιο να ορίζει τις προτεραιότητες και πάντοτε ζητούνται τα κονδύλια από τα κρατημέλη. Εγώ ως Γερμανός ε, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να βρίσκονται οι Γερμανοί πολιτικοί σε μια ιδιάζουσα θέση όταν χρειάζεται να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια γιατί πρέπει να σταθεροποιηθούν οι ποσοστώσεις στο γάλα ή γιατί πρέπει να ενισχυθεί το Ταμείο για τους μετανάστες. Ίσως πρέπει να ενημερώσουμε κάποια επιστολή των Υπουργών Ανάπτυξης ότι υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί μπορεί να μην το έχει παρήδηση. Πάση περιπτώσει όμως οι πολιτικές προϋποθέσεις ορίζονται από το Συμβούλιο το τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από εκεί και πέρα πρέπει να, υπάρξει, να δοθεί και η απάντηση του πώς θα πληρωθούν αυτές οι πολιτικές επιλογές. και τη διαδικασία με την οποία θα ρυθίσουμε τα θέματα του προπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι για το 2016 ε, μας προσφέρει ο προπολογισμό την ευκαιρία να πούμε για ποια ζητήματα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια ζητήματα έχει δεσμευτό Συμβούλιο, γιατί την το του 2020, για τις ε, πολυετής αποφάσεις που χρειάζονται και την ε, οικονομική πλαισίωση πέραν των πολιτικών αποφάσεων με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει σε απαιτήσει που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό να διεκδικήσουμε την πληρωμή να δούμε πώς έχουν ληφθεί αποφάσεις και εάν το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να τις υλοποιήσει ή εάν πρόκειται όπως το παρελθόν να δούμε μια πολιτική και υπογραμμίζω πολιτική αλλαγή στάσης σε σχέση με το Συμβούλιο. Πρέπει να δούμε εάν πέραν των δηλώσεων ε, για προγράμματα και σχέδια πίσω από αυτές τις δηλώσεις υπάρχουν και πολιτικές επιλογές. Πρέπει να δούμε τα ζητήματα της μετανάστευσης. Πρέπει να δούμε τις συζητήσεις για την περικοπή του προπολογισμού που όμως δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα όπως άλλωστε δεν λύσει και το 2015 κανένα πρόβλημα η επιλογή των περικοπών. Έτσι λοιπόν τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής που ασφαλώς θα, μας, ε, θα βρούμε μπροστά μας και το 2016 όπως και το 2015 πρέπει να έχουμε επαρκή κονδύλια για να τα αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα βέβαια είναι η κρίση των πληρωμών. Αγαπητοί συνέλφοι, η Επιτροπή μας νομίζω πάντοτε διαπίστωνε και διαπίστωσε ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο και στάση σε σχέση με τα θεσμικά όργανα. Μπορεί εγώ να είμαι κάπως πιο κοινικός, αλλά θα πω το εξής ότι εάν το Συμβούλιο δεν αποδείξει τις επιλογές σχέση με τον προϋπολογισμό του 2016 και ότι όντως εννοεί τις αναλήψεις των υποχρεώσεων να τις συνοδεύσει και από αντίστοιχα ποσά για τις πληρωμές. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε για σοβαρή πολιτική και για πράξεις. Θα μείνουμε μόνο στα λόγια του Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Έξι ακόμα ζητούν το λόγο. Δεν θα με ενοχλούσε να μιλήσετε και σύντομα δηλαδή. Κύριε Ντονάνο. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φερνάντες για την έκθεσή του και κυρίως γιατί άκουσε τη γνώμη και των άλλων επιτροπών. Εγώ ήμουν ε, ο συντάξης νομοδότης της Επιτροπής Γεωργίας και μας άκουσε. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Επίσης ε, συμμερίζομαι τις ε, προτεραιότητες για τις επενδύσεις, την απασχόληση, την νεότητα, το επιχειρήν κλπ. Και μια και μιλάμε για τον τρομερή διάλογο, θα πρέπει να δώσουμε μια αυστηρή και πολύ απτή εντολή όπως έγινε και πέρσι, έτσι και φέτος θα πρέπει να διατηρήσουμε τις θέσεις μας. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Γιατί ε, μας λέει το Συμβούλιο έχουμε πολλές ιδέες αλλά λίγα λεφτά και όχι πολύ καλές προθέσεις, όχι και πολλές προθέσεις. Ε, πρέπει για τη χρησιμοποίηση των περιθώριων, για την ανάγκη ενθάρρυνσης της έρευνας και ε, λυπάμαι που το ίτερ φαίνεται να ε, έχει μειωμένο προϋπολογισμό, ε, την, το μηχανισμό ε, συνδέοντας την Ευρώπη για το θέμα της ε, γεωργία, καθώς επίσης και για τα πιλωτικά σχέδια γιατί είναι αυτά τα οποία δημιουργούν μέλλον σε όλα αυτά πρέπει να επιμείνουμε και μετά βέβαια έχουμε και το θέμα των ιδίων πόρων και των, των εσόδων αλλά εντάξει δεν είναι τη στιγμή πριν δώσω το λόγο στην κυρία Χαουτάλα να σας πω ότι έχουμε διαρμία μέχρι τις 8 αν θέλετε να ψηφίσουμε με διαρμηνία, ε, λάβετε το υπόψη σας προκειμένου να είστε πολύ σύντομοι. Κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τους πράσινους. Μόνο εγώ θα λάβω το λόγο. Οπότε σε έχω το χρόνο. Συγχαρητήρια. Όμως στον εισηγητή πρώτα πρώτα για το αξιόλογο έργο του και πρόκειται να πούμε τις παρατηρήσεις μας αργότερα. Τώρα Δύο λόγια για την Επιτροπή που θεωρούμε ότι τώρα έχει βλάβει τη σωστή πορεία όσον αφορά το πρασίνισμα του προπολογισμού γιατί θέλουμε αυτό να γίνει και με επιταχυνόμενο ρυθμό. Τώρα όσον αφορά τις πληρωμές είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι τώρα το Global Euro πάει καλά ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές και αυτό θα έπρεπε να σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει στα σοβαρά το ζήτημα των πληρωμών. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι έχουμε εξωτερικές δράσεις και εκεί δεν υπάρχει κάλυψη, υπάρχει στέρηση ε, των πληρωμών και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ιδίως ε, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια τώρα για την μετανάστευση. Είναι απαράδεκτο ο προπολογισμό τη ε, Frontex και τη Europol να είναι τέτοια προτεραιότητα. δεν υπάρχει εντολή για έρευνα και διάσωση όσον αφορά την κρίση στη Μεσόγειο. Γιατί λοιπόν υπό αυτέ τι είναι τόσο ψηλή προτεραιότητα η Frontex. Σχεδόν διπλασιάζεται ο προπολογισμό τη υπηρεσία. Την άλλη Θα πρέπει να βοηθήσουμε την υπηρεσία ασύλου που είναι πολύ σημαντική. Δεν βλέπουμε αυτό να συνάδει με την μεταχείριση που έχει η Frontex, αλλά θα πρέπει εδώ να γίνει διόρθωση. Ήτερ. Έχουμε πει πολλά χρόνια ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι βιώσιμο και ε, διαπιστώνουμε όλο ένα και περισσότερο ότι το αναφερμένο χρονοδιάγραμμα εν ώψη του 2020 ε, δεν θα καταλήξει πουθενά. Οπότε είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι νόημα έχει τώρα έχετε πρόσθεση δύο προπολογισμό πάντω για τι διαπραγματεύσει. Ε, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τι ε, ε, τις ε, συνέπειες της έρευνας για το περιβάλλον ε, κλπ. Τώρα όσον αφορά τι εξωτερικέ δράσει. να σα αναφέρω ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει το 0,7 του ΑΕΠ για την αυρισσιακή βοήθεια ανάμεσα στο 2030. Άρα δεν θα μπορέσουμε να συγχρηματοδοτήσουμε αυτούς τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Επόμενος. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συμφωνήσω με την ανάλυση του κυρίου Φερνάντες. Θα διαπιστώσετε ασφαλώς ότι τα επιτόκια σε σχέση με την καθυστέρηση των πληρωμών ήταν σχετικά χαμηλά. Από την ε, εμπειρία μου στην ε, προηγούμενη θητεία μου σε τοπικές αρχές ε, ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και έχω ρωτήσει την κυρία Γεωργίευα την Επιτροπό εάν υπάρχει ζήτημα να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Καλό θα είναι λοιπόν να δούμε και την ανάλυση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη κατάσταση. Τι είδου συνέπειε υπήρξαν για εκείνου οι οποίοι δεν εισέπραξαν τι πληρωμέ μας. Ίσως τώρα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ίσως σε τέσσερα χρόνια να βρούμε μπροστά μας τα ίδια προβλήματα. Όπως πέρσι δηλαδή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή να αναλάβει από πλευράς της δράση και αντίδραση. Ευχαριστώ κύριος Πλένκοβιτς. Euh, Ευχαριστώ Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον γενικό εισηγητή, τον αγαπητό συνάδελφο Φερνάντε. Για τόσο έχει κάνει για να προετοιμαστεί η εντολή για το Ιντερμέρι Διάλογο του 2016. Ε, ό,τι βλέπω, ήθελε πραγματικά κάτι να κάνει. Να βρει την ισορροπία δηλαδή μεταξύ αυτών που είναι υπέρ τη ε, θέση τη Επιτροπή και αυτών που είναι υπέρ τη ε, παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, είναι νομική υποχρέωσή μα σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο δέσμευση από πριν. Οπότε η χώρα μου είναι η τελευταία χώρα που προσεχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε περιμένω το προβληματικό αποτέλεσμα του προπολογισμού 2016 για τη διαπιστώνω στις ε, προτάσεις του Ζωζέ Μανουέλ ότι ήδη έχει κατά νου την αναθεώρηση του πολιτού Δημοσιοβουλίου για το 2016. πολλέ προσδοκίε σχετικά με αυτό που ανέφεραν συνάδελφοι την πολιτική συνοχή, αλλά επίση και την πολιτική απασχολήση των νέων την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά είναι προτεραιότητες. Οπότε όσον αφορά την εξωτερική αλληλεγγύη, πήγα στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στην Μέση Ανατολή και θα πρέπει να σας πω ότι οι εταίροι μας εκεί έχουν και αυτοί πάρα πολλές προσδοκίες και παίζεται λοιπόν η αξιοπιστία ε, σε παγκόσμιο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι το πρόγραμμα Global Europe και με τον πρόεδρο της Επιτροπής μας πήγαμε στην Ουκρανία πριν μερικές εβδομάδες. Είναι πολύ ικανοποιημένη η Ουκρανία ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με την κατάληψη της χώρας και ο εθνικός προπολογισμό θα πρέπει να βρίσκεται σε ε, κατάσταση να αντέξει την κρίση. Τώρα να δούμε τι γίνεται ε, με την μετανάστευση, με την απειλή στην Μεσόγειο. Εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια αύξηση, μια αύξηση που να καλύψει καλύτερα τις ε, ανάγκες. Όπως είπε και ο θα πρέπει κάτι να εξοικονομήσουμε, μια και υπάρχει μεγάλη πίεση επί της ε, Ιταλίας τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε μια σωστή βάση για τις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν τον ε, Ιούλιο και για άλλη μια φορά μπράβο στον Ζωζέ Μανώ. Ε, ε, θα αποσύρω το αίτημά μου να μιλήσω, να πω μόνο ένα πράγμα. Το βλέπουμε και στην έκθεση του κ. Φερνάντες και στις παρεμβάσεις ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ταχύτατα η εργασία για την αθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου χωρίς μικρόφωνο. Ε, ε, εν συντομία, Πρόεδρε. Ε, θα συγχαρώ τον κύριο Φερνάντες και δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί ο συνάδελφός μου δίπλα μου το έκανε με πολλές λεπτομέρειες. Να πω το εξή μόνο. Στο σημείο 12 για τις πληρωμές. Ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρό. Βλέπω τι λέει το κείμενο πως ε, το ύψος των ε, καθυστερήσεων ε, θα είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016. Στον, στον τριμερή διάλογο είχα θέσει το ερώτημα στην κυρία Γεωργίεβα, παρουσία του Συμβουλίου. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια είχα ρωτήσει συμπεριλαμβάνουν τα πάντα ή μόνο το Ταμείο Συνοχής. Και η Επίτροπος είχε πει ότι δεν πρόκειται μόνο για τα Ταμείο Συνοχής αλλά για όλα μαζί. Όλες μαζί τις καθυστερούμενες πληρωμές. Συνεπώς, ίσως καλύτερα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε αυτό το κείμενο γιατί το κείμενο αναφέρεται μόνο στο Ταμείο Συνεχής. Ε, θα κάνω και μια πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Τελειώσω ότι 21 δισεκατομμύρια ε, δεν δεσμεύτηκαν το 2014 θα βοηθήσει την εκαθάριση ε, των καθυστερούμενων πληρωμών τουλάχιστον το 2016. Αλλά ε, ποιος ξέρει τι θα γίνει το 2017, 2018, 2019 και 2020. Γιατί εκεί θα επανέλθουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα. Οπότε ή θα μειώσουμε την ανάληψη ε, υποχρεώσεων ή θα αυξήσουμε τις πιστώσεις πληρωμών. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Κομισιόν ενδεχομένω θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το λεγόμενο backlog, το αναμενόμενο δηλαδή ε, ποσό ανεξόφλητων λογαριασμών είναι στα 2 δισεκατομμύρια για τα προγράμματα 2007-2014. Αυτό συστήθηκε δηλαδή με ιδιαίτερη τα τελευταία χρόνια. Για τα νέα προγράμματα 2014-2020 πολιτικής συνοχής όπου ιδιαίτερα έχουμε το ποσοστό των ε, ραλ των συνολικών ραλ, τα 2 τρίτα των συνολικών ραλ δηλαδή όπου καθυστερούν ε, οι εξοφλήσεις των προγραμμάτων θα έχουμε κάποια ποσά λογαριασμών προς τα τέλη του 2016 κάποια μάλιστα και στην τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2016 που θα μείνουν ανεξόφλητες, ε, ανεξόφλητα τα τιμολόγια διότι πρέπει να γίνει ο έλεγχός τους, ε, να εξεταστεί ότι όλα έχουν τηρηθεί όπως πρέπει και λοιπά. θα μπορούσαν να πληρωθούν εγκαίρως. Ίσως να υπάρξουν και κάποιες μικροδιακοπές ή άρσεις πληρωμών ώστε να γίνει η αρσεις πληρωμου ωστε να γινει η επαληθευση του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα χρόνια και επιπλέον αναμένεται ποσότητα κάποιων ε, τιμολογίων που δεν θα εξοφληθούν που όμως θα είναι πάρα πολύ λίγα και σε ποσά σε σχέση με αυτά που μένουν στο τίτλο 1β γιατί δεν έχουμε backload επί παραδείγματι για την γεωργία στον, στους κύριους ε, τομείς της, στις ούτε και στις διοικητικές δαπάνες αυτά εν γέννη λοιπόν τα δύο δις που ανέφερε και η Αντιπρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια αφορούν τα προγράμματα 2007-2014. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Φερνάντες, για να ολοκληρώνουμε. Και διευκρινίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 6 το βράδυ. Λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων ανάμεσα στη δημοσίευση του σχεδίου και τις ολομέλειες του Ιουλίου τροπολογίες μπορείτε να καταθέσετε μόνο στα αγγλικά και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται να γίνει στις 23 Ιουνίου όπως είπα, στενά χρονικά περιθώρια. Ψηφίζουμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. 14 Ιουλίου αρχίζει ο τριμερής διάλογος. Κύριε Φερνάνδες. Όλοι θέλουμε να μην ε, επικρατήσει ε, η συζήτηση για τον τριμερίδα λόγω των πληρωμών στον προπολογισμό του 2016 να μην τον επισκιάσει θα λέγαμε έχει ήδη γίνει τόση συζήτηση και από την Επιτροπή και σε εμά. για τη συζήτηση λοιπόν την περαιτέρω έχετε κάτι να μας προσθέσετε προτεραιότητες Φερρυπίν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες νομίζω ότι είναι σαφή το πρώτο κομμάτι του εγγράφου της ε, προσχεδίου εκθεσής μου, νομίζω καταγράφονται. Μίλησα ήδη για αυτούς τους στόχους, για αυτές τις προτεραιότητες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αδέρφους ε, ε, για τα καλά τους λόγια και για τη στήριξη που μου παρήσχαν. Περιμένω τις ε, προτάσεις τροπολογίας, τροπολογιών τους. Από ό,τι φαίνεται οι προτεραιότητες που έχουμε συμπεριλάβει είναι καλές, ε, είναι καλές και οι προτεραιότητες οι οποίες είπε η Κομισιόν. Ε, θα συνεχίσουμε την εργασία μας και βλέπω ότι επικρατεί μια ατμόσφαιρα ενωτική και αυτό είναι πολύ καλό στην Επιτροπή μας. Ασφαλώς και υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Ε, δεν είναι δυνατόν οι προτεραιότητες και οι δεσμεύσεις να μειωθούν, να μειώνονται. Το πολιετές δημοσιοκοπλαίσιο πλαίσιο ε, το οποίο διαθέτουμε εγκρίθηκε με ομοφωνία στο Συμβούλιο. Τώρα δεν είναι δυνατόν το Συμβούλιο να αμφισβητήσει αυτό που υιοθέτησε με ομοφωνία. Πώς να το δεχτούμε αυτό οι δεσμές που έχει αναλάβει το Συμβούλιο είναι σαφείς, η ευελιξία είναι σαφής, οι πολιτικές προτεραιότητες ε, τις οποίες υποστηρίζουμε νομίζω ότι υποστηρίζονται τουλάχιστον δημοσίως και από το Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε λέω με αυτή τη δουλειά και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό Υπάρχει βέβαια και άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα προσθεθεί στη συζήτηση μέχρι το 2020 είναι ο ορίζοντας 2020 και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός συνέοντας στην Ευρώπη δύο προγράμματα τα οποία, στα οποία θα πρέπει να επιστρέψουμε τα ποσά τα οποία τους έχουμε αφαιρέσει. Εμείς μιλάμε για ε, ε ανασκόπηση και αναθεώρηση του προπολογισμού, του δημοσιονομικού πλαισίου και ελπίζω και η Κομισιόν να μιλήσει για το ίδιο πράγμα. Το Συμβούλιο δεν μιλάει για τίποτα. Αλλά όταν μιλάει συνήθως μιλάει για την ανασκόπηση και όχι για την ε, ε, μεταρρύθμιση. Ε, πάντως ε, ο προπολογισμό θα πρέπει να σέβεται τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις μας. Πρόεδρος, ελπίζω ότι ε, θα ε, καταφέρουμε το Συμβούλιο να λάβει δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Περνάμε σημείο 4. Κινητοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Δίνω το λόγο στον κύριο Σαβάρμα. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να σας τα πω στα αγγλικά, ως συνήθως. εφαρμογή από την Φιλανδία και όλα είναι πάρα πολύ απλά εκτός από ένα θεματάκι το οποίο θα σου το εξηγήσω. Ε, αφορά με την ε, Broadcom μια εταιρεία που έκλεισε στην Φιλανδία και αυτή η εφαρμογή αφορά 500-868 εργαζομένους ε, οι οποίοι απολύθηκαν ως ε, πλεονάζοντες ως υπεράρθμοι τέλο πάντων και είπαμε ότι τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε αυτές τις ε, απολύσεις της ε, Broadcom και ε, να κλείσει δηλαδή το εργοστάσιο τελείως συνέβη το εξή. Είπαμε ότι το έκανε αυτό η κυβέρνηση ούτως ώστε να γίνουν καλύτερες διαφορετικές αλλαγές. Κάτι το οποίο βέβαια το συναντούμε ως στοιχείο σε όλες τις εφαρμογές περιπτώσει εφαρμογής τέλο πάντων αυτού του κανονισμού. Οπότε δεσμευόμαστε 100% από τον κανονισμό και το γράμμα του νομοθετή μας οπότε και εγώ θα πρέπει να κατεβάσω μια τροπολογία ε, σε πλαίσια του σχεδίου έκθεσης μια μικρή αλλαγή του κειμένου και θα λέω ότι θα πρέπει να είμαστε τίμοι, ειλικρινείς όσον αφορά τη δράση μας Να πούμε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο συνέβη μόνο ε, στην παγκοσμιοποίηση, αυτό δεν είναι ειλικρινέ. Οπότε θα προτείνω αυτή την ελαφρά αλλαγή του κειμένου σε αυτό το κείμενο και ελπίζω θα το εγκρίνει η, Ευρώπη η Επιτροπή μα και θα προσθέσουμε ότι αυτέ οι απολύσει τη Botcom εν μέρη οφείλονται στην αλλαγή αυτή τη τάση αυτή τη στροφή αυτού του κλάδου τη φυλακή οικονομία ακριβώς όπως και η Νόκια έκανε το 2011 και θα καταλήγουμε το ότι αυτά τα γεγονότα συνδέονται ε, ουσιαστικά και άμεσα με την παγκοσμιοποίηση κλπ. κλπ, λοιπά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρά το ότι αυτό το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση ε, ελαφρύνει κάποιο, κλείνει κάπως τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης, δεν μπορούμε να πούμε στο κείμενό μας ότι δεν υπάρχει και, και η αγορά η ΝΟ και κάνει κάποια στρατηγικά ασφάλματα επί ετών. Οπότε τελικά περί αυτών των σφαλμάτων πρόκειται και όχι περί κάποιου φανταστικού μαγικού ε, πλάσματος όπως είναι η παγκοσμιοποίηση. Οπότε αυτά θα προτείνω και κατά τα άλλα όπως σας είπα είναι απλό το ζήτημα και μια που είναι 8 και το δεν σας πω άλλο. Merci, M. Sarvama. Κύριε Σαρβάμα, σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος. Ναι, έτσι συμβαίνει η παγκοσμιοποίηση. Και για να είναι κάποιο επιλέξιμο για να καλυφθεί από αυτό το ταμείο τη παγκοσμιοποίηση, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πώς, αποφασίστηκαν αυτέ οι απολύσεις κατά πόσο πραγματικά συνδέεται με το πρόβλημα Γιατί σε άλλε περιπτώσει είναι θέμα διαχείριση των επιχειρήσεων, είναι θέμα των, των μάλλον ακολουθηθισών στρατηγικών. Δεν θέλει κανεί το λόγο από ό,τι βλέπω. Ε, διευκρινίζω ότι οι τροπολογίε θα μεταθούν μέχρι τι 16 Ιουνίου στι 4 η ώρα. Θα συζητήσουμε στι 23 Ιουνίου και το θέμα θα κατέβει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Τώρα, όσον αφορά την ψηφοφορία. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική κάρτα. Τοποθετήστε την στη συσκευή. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για την τεχνική αρρωγή όσον αφορά την έκθεση Ζωαλ Ντεπρέ. ΤΑΦ Α2015. Πρώτη διάταξη υπέρ ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία. Δεύτερη παραγωγή τροπολογία υπερθυμών 3 υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 2, τροπολογία 4, υπέρ ο συγκητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευσα. Le scrutin est ouvert. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίπτω την τροπολογία. Παραγωγός 2. Τροπολογία 5 υπέρ. Ο ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. το Τροπολογία 6 υπέρ. Ο συγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Το Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Υπέρ ο Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2 2Γ, τροπολογία 8, υπέρ. Ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 9, υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ξεφύρουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγραφός 4. Α. Κατά ο εισηγητής. Πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 4. Τροπολογία 11. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρα. κατά επαλήθευση ψηφίζουμε τροπολογία 11 Ναι, ψηφίσατε, αλλά δεν με βέβαιος να διαμορφώθηκε πιο ψηφία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό κάνουμε επαλήθευση και ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας. εγκρίνεται. 19-16. Παράγραφο 4, τροπολογία 12. Υπέρ ο Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 4 έχουμε τροπολογία 13. Κατά ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 β. Τροπολογία 14. Υπέρ ο υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 16-15. Παραγραφός 5, τροπολογία 15. Κατά ο Ζήγητος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 6, τροπολογία 16 υπέρ ο υπερ υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6α, τροπολογία 17, κατά ο υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 6 β. Τροπολογία 18 υπέρ ο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 γάμα 19 περ κατά αποχές εγκρίνεται 7α τροπολογία 20 υπέρωση, ο ποινή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι επαλήθευση Πρόκειται για την τροπολογία 20. Τέλος. Εγκλίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 21, κατά, ο εισηγητής. Τίποτα, έχουμε προφορική τροπολογία. λέει τώρα η φράση τονίζει τη σημασία, τονίζει την σημασία. Highlight the importance. Κατά σου έχετε υπέρ, κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζουν. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τρώγει παράγραφος 8, το πρωί 1 υπέρ ο υπέρ, κατά, επελήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας που δεν ψήφισε. Πέρασε. Εγκρίνεται το κείμενο 27, 5 και 3 αποχές. Κύριε Γκαντιθάπολη, κύριε τη μεταφορά πιστώσεων. Ονομαστική ψηφοφορία. Συγκεκριμένη τη μεταφορά πιστώσεων που αφορά την εκαθάριση. Ψηφίζουμε το κείμενο. υπερος Υπέρος Σκοτάει του που δεν Εψήφισαν όλοι. Όχι. Εντάξει. Πέρας. 27. 3. Τρεις εποχές. να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χόλμαγερ για τα άλλα τμήματα. Έχουμε και άλλη μια έκθεση, η οποία όμως ε, διαβιβάστηκε ε, αργά. Το σε 5 για το σε 3. Κυρία Χόλμαγερ. Καταρχάς, πρώτη μεταφορά αφορά στήματα προσωπικού. Έχω μια σαφή παράκληση να μην γίνονται οι προτάσεις δύο ώρες πριν από τη συνεδρίαση για να μπορούμε να τις μελετούμε πολύ πιο σοβαρά. Έχουμε τους συμβασιούχους, contract agents, που δεν μπορούν να πληρωθούν εάν δεν ενισχυθεί ο προϋπολογισμός αναλόγως, γιατί ήταν τέτοιες σημαντικές οι περικοπές του προηγούμενου έτους που δεν αρκούν ε, τα ποσά για να τους Έχουμε λοιπόν 594 από τα allowances που μπορούμε να πάρουμε και 0,9 επίσης, οπότε έχουμε συνολικά 4,6 για το λοιπόν προσωπικό. Παρακαλώ να το εγκρίνουμε. Ο πρόεδρος. Σε τρία. Ασφάλεια. Συμφωνείτε για τις πιστώσεις αυτές κυρία Χολμάιερ του ΣΕΤΡΙΑ. Ε, πρόεδρε, το προσωπικό ήμασταν τώρα. Χρειάζονται τρει ψηφοφορίε. Η μία είναι το προσωπικό, η άλλη η ασφάλεια και μετά το EU Lisa. Καλώ. Σε πέντε πρώτα. Παρακαλώ. Ε, ναι, το είπε η συγγετρία. Δεν είναι φυσιολογικό να ψηφίσουμε μια μεταφορά πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ με πληροφορίες που έφτασαν τελευταία στιγμή και είναι ελλειπείς. Ε, είναι σημαντικό αυτό το ποσό, αλλά και ακόμη και αν δεν ήταν τόσο σημαντικό, δεν είναι σωστός τρόπος αυτός. Ασφαλώς δεν αποτελεί αυτό που λέω κριτική στην συγγήτρια, αλλά δεν το βρίσκω φυσιολογικό και λογικό. Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Έχουμε και άλλη μια περίπτωση αργότερα, και το λέω από τώρα, για να μην παρέμβω αργότερα, το θέμα με το, το EU Λάβαμε την πρόταση σήμερα στις 6 το απόγευμα. Και πάλι δεν επικρίνω την συγγήτρια γιατί ξέρω ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της. Αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάνουν πληροφορίες τόσο καθυστερημένα. Θα ήθελα να αναβάλουμε την ψηφοφορία ε, στο μέτρο του δυνατού γιατί αλλιώς εμείς θα απόσχουμε ως ο πολιτική ομάδα. Κυρία ε, ε, βέβαια δεν σοβαρή διοίκηση όταν ε, δύο ώρες ή αν ούτε μια ώρα πριν από την έναρξη μας ε, κάνει τις αιτήσει. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Ε, Διερωτώ με πάντως τι κάνει Για να ουτε μια ωρα πριν απο την εναρξη μας κανει τι αιτησει ναι συμφωνω απολυτως διερωτω με παντως τι κανει η επιτροπη και το Κοινοβούλιο όταν χρειάζεται τόσες εβδομάδες να πηγαίνει ένα φάκελος από το ένα επιτελείο στο άλλο για να εγκριθεί και να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε το προσωπικό μας. Εν πάση περιπτώσει εκφράζω την οργή μου ξεκάθαρα για την κατάσταση αυτή διότι χρειάστηκε να πάει μπαλάκι πινκ πονγκ από το ένα επιτελείο στο άλλο για να φτάσουμε τώρα να λέμε πρέπει να δώσουμε την, ε, τα επιπλέον ποσά γιατί αλλιώς δεν έχουμε πληρώσει πληρώσουμε το προσωπικό. Το μόνο που με κάνει να, το, να συμφωνώ είναι γιατί ξέρω τι είναι το διακύβευμα. Αλλά συμφωνώ 100% με την Αλφαέντερ. Πού είναι ο αρμόδιος διευθυντής? Ίσως θα ήταν καλό να μας εξηγήσει ένα λεπτάκι. Γιατί τα έχει ακούσει από μένα, ναι, είδε. Έτερος. Ο διευθυντής. Εκ μέρους της Επιτροπής. Του Κοινοβουλίου. Πώς καταντήσαμε σε αυτά τα χάλια κύριε Ρίφιντα. Υπήρξαν κάποιες προ... προβλέψεις. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο να σας εξηγήσω. Η κατανομή αυτού του ποσού 2,25 εκατομμύρια προβλέπονται για την συνέχιση των ψημάς υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων που προσλαμβάνονται Συνε, κύριε Χόλμα, ζητάτε το λόγο. Δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες ε, πρόσληψης προσωπικού ακολουθούν αυστηρούς κανόνες. Ε, αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις και για αυτό το λόγο οι πολιτικές ομάδες ζήτησαν πρόσθετα ποσά έτσι ώστε να γίνει σταδιακή πρόσληψη προσωπικού για τις πολιτικές ομάδες εξασφαλίζοντας μια συνεχή υπηρεσία από τις εκλογές και μετά. Γνωρίζετε το καινούριο οργανόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε από 1η 1ου 2015. Μετά έχουμε το ποσό του 1,6 εκατομμυρίου για τους επισημάς υπαλλήλους ασφαλείας, δεδομένης της σημερινής κατάστασης, επιταχύναμε αυτή τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ασφαλείας. Και τέλος, έχουμε την πολιτική ε, και μέσω αυτού του ποσού ε, προσλήθηκαν οι πάλι με αναπηρίες. Επίσης έχουμε ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό αδειών μητρότητας και πατρότητας, ε, κάτι που μας οδήγησαν στην, ε, οδήγησε στη δημιουργία προβλημάτων τα οποία τα ξεπεράσαμε. Όμως σας εξηγώ ποια είναι τα προβλήματα, είναι δύσκολο παίρνει χρόνο κάθε φορά να εξεταστεί το καθέτημα. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναβάλλετε τη για μια επόμενη συνεδρίασή σας έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος να σας ενημερώσω λεπτομερώς. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι για τις 23 Ιουνίου. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τότε. Ε, τότε να κάνω και μια ερώτηση, Ευθυντή, αν επιτρέπετε. Πώς θα γίνει όταν δεν θα έχετε πια τη δυνατότητα να πληρώνετε το προσωπικό και θα πρέπει οι ομάδες να βρουν τη λύση. Μπορεί να περιμένουμε τρεις εβδομάδες και τα λοιπά, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε ακόμη την πρόταση. Απάντηση. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στην ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι κάποιες από τις συμβάσεις θα ε, κλείνουν και πρέπει να ανανεώθουν αμέσως πριν από το καλοκαίρι. Μια ψηφοφορία λοιπόν σήμερα θα μας διευκόλυνε. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι σας εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα και αντιμετωπίζετε σοβαρή δυσκολία δηλαδή προς το να το υιοθετήσετε σήμερα και στο συγγνώμη. Καλώς λέει ο πρόεδρος, καλοκαίρι. Αλλά καλοκαίρι είναι 21 Ιουνίου και 23 Ιουνίου είναι η ψηφοφορία μας ναι αλλά η διοίκηση είναι διτεθειμένη να κάνει ό,τι γίνεται για να εξελιχθεί ομαλά όλο αυτό. Καλά, τότε θα περιμένουμε 23 Ιουνίου. Κυρία Χολμάιερ. Θα γίνει, θα γίνει απόλυση του προσωπικού αυτού ή όχι. Όχι λέει ο διευθυντής, δεν υπάρχει το ζήτημα. Απλώς μπορούμε τώρα να κάνουμε μία περιορισμένη παράταση συμβάσεων. Αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν εάν θα μείνουν μέχρι να ανανεωθεί το συμβόλαιο, τα συμβόλαιά τους, επειδή εσείς καταθέσατε καθυστερημένα τα έγγραφα. Απάντηση. Όχι, τα έγγραφα χρειάστηκε να διορθωθούν σε ένα τομέα, ως εκ τούτου προέκυψαν οι καθυστερήσεις. Ο πρόεδρος θα τα προτιμώσουμε όλα και υποθέτουμε όλοι ε, στις 23 Ιουνίου θα είναι υπέρ, θετική τέλο πάντων, οπότε θα είναι όλα έτοιμα προ εκείνες. Δεν πρέπει. Ναι, καταλαβαίνω ποιε είναι οι επιφυλάξει σχετικά με αυτό, αλλά υπάρχει κάποια πιθανότητα μέσα σε ένα 15 μέρο αυτό το ποσό να μεταβληθεί. εχει γίνει και η ελάχιστη συζήτηση ε, όσον αφορά τι θα γίνει. Και αν δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο, εντάξει. Αν δεν υπάρχει επομένω ε, κάποιο κίνδυνο να αλλάξει αυτό το ποσό μέσα σε ένα και αν αυτή, αυτό το, το αίτημα για την πίστοση είναι θεμητό, γιατί να μην ψηφίσουμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό έφτασε τελευταία στιγμή και αυτό ενοχλεί, αλλά είναι πρόβλημα. Εκτός μικροφωνού ο Πρόεδρος. Συμφωνώ σε ένα σημείο με τον συνελφό Ντεπρέ ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ουσία, ως προς το περιεχόμενο. Είναι σαφής η κατάσταση. Το θέμα είναι ο τύπος και να έχει την ασφάλεια το προσωπικό. Δεν θέλω να τους ε, προξενήσουμε δυσκολίες ή ανασφάλεια. Αλλά επικρίνω το γεγονό ότι δεν κατατέθηκαν εγκαίρω τα σχετικά έγγραφα. Αυτό θέλω να τονίσω. Μου φαίνεται ότι η κατάσταση είναι αρκετά στριμωγμένη. Λίγες ώρε. πριν πρέπει να διπηρεθεί ένα θέμα να έρχεται το έγγραφο. Δεν είναι καλό. Και σε μια ολομέλεια στο Στασβούργο είμαστε εμεί στο ημικύκλιο κάποια ώρα, οπότε δεν μπορούμε καν έστω και τη στιγμή να μελετήσουμε το έγγραφο. Νομίζω ότι αυτό είναι τραγική έλλειψη επικοινωνίας. Αν πρέπει κάποιος να στείλει το έγγραφο τόσο αργά, γιατί να μην έχει διαβαστεί το έγγραφο εγκαίρως. Ε, όπως να ξέρουμε πότε θα έρθει. Δεν βρέθηκαμε σε αυτή τη θέση. Θα πρέπει να το έχουν πει αυτό στην εισηγήτρια. Έγκαιρ ότι έτσι θα γίνει. Για κοιτάξτε, ποιος είναι ο υπεύθυνο υπάλληλο και ας αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία σχετικά. Μπέγκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, ε, καταλαβαίνουμε αυτά που λέει ο Σάνφος Αφετέρου, Πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε και έχω εγώ παρελθόν εδώ σε αυτήν την επιτροπή να τηρεί και η διοίκηση τις προθεσμίες για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Όσο λοιπόν παραγνωρίζουμε αυτή τη διάσταση και όσο αφήνουμε χαλαρά τα χαλάρια χάνουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες και να μπορούμε εμείς, η Επιτροπή ή ο εισηγητής, να ενημερωνόμαστε εγκαίρως ή δάλλως θα πρέπει να ε, σκεφτούμε άλλες ε, άλλη συμπεριφορά και άλλες δράσεις αντί της διοίκησης, όχι βέβαια των συνεργατών υπαλλήλων, αλλά των, εκείνων που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις καταστάσεις. Ο Πρόεδρος, ε, ας ψηφίσουμε πια. ας διαφώτισε αρκετά η Επιτροπή. Μας είπε η συγκήτρια ότι διαμαρτύρεται ότι είναι παράδεκτη κατάσταση, δεν πρέπει να επαναληφθεί, αλλά ότι υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν σε δυσκολία οι υπάλληλοι, οι πολιτικές ομάδες, η γραμματεία και ως εκ τούτου θα πρέπει να δεχθούμε να ψηφίσουμε. το του λεχθέντος και μια και πρόκειται για μεταφορά πρέπει να γίνει ονομαστική η ψηφοφορία και αρχίζει τώρα. voyez. Le scrutin est clos. Et le dispositif. αποχής και ψήφοι υπέρ ε, ισοδύναμες, αυτό δείχνει ακριβώς την διάθεσή μας. Για το ΣΕ3 κυρία Χολμάιερ, ε, μεταφορέ πιστώσεων και υλοποίηση, αναβολή, τι έχετε να μας πείτε. Δεύτερο σημείο λοιπόν, ασφάλεια. 7 εκατομμύρια. Υποστηρίζω την εντολή. Ε, έχει να κάνει με το επεισόδιο εκείνο όταν Κούρδοι διαδηλωτές ε, εφόρμησαν στο κοινοβούλιο. Άλλοι ιδιαίτερα άλλη αιτία ιδιαίτερα έχει να κάνει με την περίοδο μετά τις επιθέσεις κατά του Σαρλί Επδό και την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ε, ασφαλείας στο Κοινοβούλιο έχουν γίνει εντατικά μελέτες της κατάστασης και για τις εισόδους που θέλουμε να μείνουν μένα ανοιχτέ και διαφανεί κτλ. Αλλά από την άλλη θέλουμε και δεν είναι ασφαλεί. Επομένω, μιλούμε για τζάμια ασφαλείας και επιπλέον ελέγχους και στάδια στην είσοδο. 7 εκατομμύρια όπως σας είπα η μεταφορά για τον εξοπλισμό από το αποθεματικό έκτακτων αναγκών και θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα, ο, τουλάχιστον οι συγκητές, όταν θα έχουμε ακριβέστερα στοιχεία από το Κοινοβούλιο. Κατά τα άλλα το υποστηρίζουμε. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Μάλλον ψηφίζεται n'avez pas tous voté. Εντάξει τώρα. Πέρασε ψηφοφορία. Σημαντική πλειονοψηφία υπέρ. Η υλοποίηση, κυρία Χολμαϊρ. Και κτίρια. Τελευταίο σημείο, ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα αυτό των κτηρίων που κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια. Με την κυρία Χόφμαν έχω συζητήσει το θέμα αυτό εντατικά. Η Επιτροπή, και αυτή είναι απερίφραστη κριτική την οποία καταγράφεται σε μια γνωμοδότηση, δεν ε, ενθάρρυνε την υπηρεσία να μας καταθέσει τα έγγραφα που χρειαζόταν. Στις 4 το απόγευμα σήμερα λοιπόν μόνο μπόρεσα να δω τα έγγραφα 200 σελίδες φάκελος και πρέπει να πω ότι δεν είμαι και τόσο ε, ειδική στα θέματα του γαλλικού οικοδομικού δικαίου. Εν πάση περιπτώσει πέραν των 200 σελίδων του εγγράφου υπάρχουν χιλιάδες ακόμα σελίδες με σχέδια, με ε, αρχιτεκτονικά σχέδια κτλ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τώρα τι δεν περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Πρέπει να πω και πρέπει να πω ξεκάθαρα για τα πρακτικά ότι μια και έχουμε να κάνουμε με κόστος προγραμματισμού, το κόστος προγραμματισμού πρέπει να εγγράφεται στο συνολικό κόστος του έργου. Δεν μου είχε κοινοποιηθεί νωρίτερα, τώρα το βλέπω. Σε σχέση με το κόστος λοιπόν έχουμε πρώτη φάση 10,2, 11,3 στη δεύτερη φάση, 21,5 στη συνέχεια με μια μεγάλη επιχείρηση γενικά και έχουμε την διάθεση που εκφράζεται για αποδοχή της κοινοποίηση με 30.000 που θα δεχθούμε αλλά δεν θα δεχθούμε το αίτημα της υπηρεσίας για 2 εκατομμύρια αποθεματικό ασφαλείας. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν μπορώ να δώσω ένα-δύο εκατομμύρια με ερωτηματικό μόνο. Πρέπει να έχουμε πιο προσεκτικό προγραμματισμό. Διατυπώνω λοιπόν και μια γνωμοδότηση μαζί με την κυρία Χόφμαν, στην οποία καταγράφουμε όλα τα ποσά και όπου λέμε συγκεκριμένα, απευθυνόμενοι προς την Επιτροπή, ότι μια υπηρεσία να έχει έναν, ε, ένα σχεδιασμό οικονομικό και για τα κτίρια με κοστολόγηση σε κάθε στάδιο και βεβαίως και εμείς έχουμε αντίστοιχες ε, διατάξεις και προσπαθούμε να κάνουμε στο δυνατόν πιο οικονομικά τα, να εκτελούμε στο δυνατόν πιο οικονομικά τα σχέδιά μας. Εν πάση περιπτώσει διατυπώνω τις επικρίσεις μου και καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να Καλή και εκείνη και να ενθαρρύνει από πλευρά της τις υπηρεσίες να μας ενημερώνουν για τις ε, πληρωμές σε κάθε λεπτομέρεια. Λαμβάνω λοιπόν πιο συγκεκριμένες ε, ε, πληροφορίες. Θέλω να ξέρω ακριβώς πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα πριν και μετά, ποια είναι τα ακριβή ποσά και εάν χρειαστεί κάποια αλλαγή θέλω δέσμευση της Επιτροπής και της υπηρεσίας ότι θα ενημερώσουν. Δεν πρόκειται να δώσουμε λευκό επιταγή δηλαδή για επιπλέον δαπάνες. Σημειώνω επίσης επικριτικά ότι δεν προβλέπονται ε, δαπάνες για ανελκυστήρα και σημειώνω ότι θέλουμε ενημέρωση για την πρόοδο του, της ανέγερσης του κτηρίου τακτικά ώστε να γνωρίζουμε επαρκώς τι προχωρεί. Το Ιουλίζα αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο σε μεγάλο βαθμό σε ε, εμπορευματοκιβώτια και όχι σε κτίρια. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε κυρίως εμείς που απαιτούμε και την ασφάλεια των δεδομένων την επαρκή κτηριακή υποστήριξη. Αλλά δεν μπορώ πέραν του ότι δέχομαι ότι πρέπει να γίνει η ανέγερση του κτηρίου δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έπρεπε τέτοια να έχουμε τόσο πρόχειρη δουλειά, τόσο περίπλοκη, τόσο χαοτική και τόσο τις τελευταίες στιγμές. Σας ευχαριστώ. Τι λέτε να αποφασίσουμε σήμερα ή να μεταθέσουμε την ψηφοφορία σε 15 μέρες μετά. Πρέπει να ρωτήσετε το ίδιο Λίσα και την Επιτροπή, γιατί είχαμε αναβάλει και την προηγούμενη φορά. Μήπω πρέπει αντί να εγκρίνουμε να δώσουμε μια τελείως αρνητική γνωμοδότηση και να στήσουμε νέα κοινοποίηση εξ αρχής. Δεν φταίω εγώ βέβαια γι' αυτό, αλλά πέραν της νομοδότησης δεν μπορούμε να προσφέρουμε και πέραν των ποσών επίσης δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα άλλο εγώ θα πρότεινα να εγκριθεί η γνωμοδότηση για να εκφράσουμε την επικριτική μας στάση, να περιορίσουμε, να ορίσουμε μάλλον την κατάσταση και τα περιθώρια και ενδεχομένως να δώσουμε ένα περιθώριο για την έγκριση νέας, ε, νέου οικοδομήματος. Le document, le draft vous a été distribué. Vous en avez pris connaissance Το έγγραφο σα διανεμήθηκε σήμερα, ε, το έχετε υπόψη σα, Προτείνω να μην ψηφίσουμε σήμερα. Πρόεδρε, ακριβώ αυτό είπα. Ότι εδώ δηλαδή, στο Στρασβούργο, έχουμε τέσσερα διαφορετικά οικόπεδα πάνω στο οποίο πρόκειται να γυρθούν κτίρια. Έχουμε ακριβή αριθμό τετραγωνικών μέτρων. Πόσα είναι τα διαθέσιμα τώρα, πόσα εμπορευματοκιβώτια υπάρχουν, τι προβλέπετε ως σχέδιο, κύριο κτίριο δηλαδή που θα ανακαινιστεί και επέκταση με δύο μικρότερα κτίρια που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ασφάλεια και την παροχή ενέργειας και πάλι με επακριβή με, ε, ε αναφορά τετραγωνικών 5.800 συγκεκριμένα. και θα έχουμε συνολικά στο τέλος 5.025 τετραγωνικά χώρο εργασίας για 166 άτομα από τα 44 που έχουμε τώρα ως προσωπικό άρα μπορεί να υπάρχει επαρκής χώρος για το προσωπικό του Λίσα ε, υπάρχει ένα ποσό 23,5 ε, ποσών χωρίς το αποθεματικό ασφαλείας, 24 μέτρα το αποθεματικό ασφαλείας, 173 εκατομμύρια θα κοστίσει το κτίριο, τα υπόλοιπα τα δίνει το υπόλοιπο του Στρασβούργου. Η ανακαίνιση 11,9 και η επέκταση 2% είναι το περιθώριο σφάλματος και 6.000 για την απομάκρυνση και καταστροφή εμπορεύματοκιβωτίων. Οι επίκρισεις μου απευθύνονται κυρίως στο Ιουλίθα αλλά και στην Επιτροπή διότι χρειάστηκε υπερβολικά μακρύ χρονικό διάστημα για να μα δώσουν τις πληροφορίες. Δεν ήταν αρκετά σαφείς και συνοπτικές και επίσης η Επιτροπή θα μπορούσε να μην ζητήσει τα χρήματα αυτά γιατί έχουν ήδη διατεθεί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα δηλαδή σχέση με το 1,2. Επικρίνω με την γνωμοδότηση μου ότι το γεγονός ότι προχώρησε έτσι η κατάσταση και η έγκαιρη προειδοποίηση ότι δεν ενημερώθηκε δηλαδή εγκαίρωση ο εισηγητής με το Ιουλίσσα 17 ή 19 εκατομμύρια που γίνανε μετά 24 και εν τέλει ζητούμε τα 2 εκατομμύρια για το αποθυματικό ασφαλείας να μην ε, προβλεφθούν με τη δυνατότητα για αύξηση κατά 15%. Θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στις δαπάνες οι οποίες έχουν προβλεφθεί τώρα και αν χρειαστεί να μας ενημερώσουν και να δώσουμε άλλη επιπλέον έγκριση. Αυτά μπορώ να κάνω από την κατάσταση που έχω μπροστά μου. Είναι γνωστό εδώ και εβδομάδε, ότι είναι ένα απαραίτητο έργο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ε, εδώ και κάποιο καιρό έχω παρατηρήσει ότι μας υποβάλλονται έγγραφα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να μελετήσουμε. Η εμπειρία μου στη ζωή είναι η εξή. Όταν κάποιο αποφασίζει για κάποιε δαπάνε, αυτέ οι δαπάνε θα πρέπει να τι γνωρίζει εκ των προτέρων και έγκαιρα. Από ό,τι φαίνεται, η γνώμη μα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν όμω έτσι έχουν τα πράγματα, τότε εξορισμού θα πρέπει να ψηφίσω κατά. Ποιο άλλο θέλει τον λόγο? Ωραία, θέτουμε σε ψηφοφορία το κείμενο τη έκθεση Χολμέγια. Ποιο είναι υπέρ? Merci, les mains, contraire. Κατά. Eh bien, je crois qu'on a une majorité pour euh, ratifier cette opinion. Εγκρίνεται. Ich kann mich nur leider entschuldigen, dass äh, spät Ich war keine Absicht. Λυπάμαι που έγινε έτσι. Δεν ήταν εκπροθέσεως μόνο σήμερα στις 4 το απόγευμα έλαβα τα στοιχεία. Καλά λέει ο Πρόεδρος, αλλά να σταματήσουν αυτά. Να κάνει επιτροπή τα δέοντα. Και δεν θα δεχόμαστε από εδώ και μπρος εκθέσεις που φτάνουν τελευταία στιγμή πριν από τη συνεδρία διότι δεν είναι διαδικασίες αυτές σωστές. Όσοι δεν είναι για τους Η διακυβέρνηση στην Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό έρχεται από τη διαδικασία. Λοιπόν, οι διαδικασίε εδώ δεν είναι ικανοποιητικέ και πρέπει να το σημειώνουμε. Και παρά τι πιέσει τη κυρία Χολμάιερ. Να αφήσουμε το ΑΕΣΠΕ για τις Βρυξέλλες. το θέμα της ασφάλειας, τα λοιπά, το αναβάλουμε, έτσι, καλά. Τελευταίο σημείο. Συζήτηση στην Επιτροπή σε 15 μέρες περίπου. Φερνάντες. Να μας πείτε τι έγινε ο τριμερής διάλογος